Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία σύντομα να ε, προσεγγίσουμε κάπως τη συζήτησή μας και τα βασικά σημεία καθώς οδεύουμε προς το τέλος της ακρόασης. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. Παλιές ιδεολογίες τύπου ε, δωρητού δικαιούχου δεν ανήκουν, δεν χωράνε στο νέο πλαίσιο θα είναι σημαντικά τα επόμενα χρόνια για να προσαρμόσουμε στις νέες πραγματικότητες ε, μια νέα εταιρική σχέση για ένα καλύτερο κόσμο. Χρειάζεται αλλαγή υποδείγματος από τους σημερινούς στόχους της χιλιετίας προς στόχους αηφόρου ανάπτυξης και είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για καλύτερη καταπολέμηση της ένδυας μέσω της ένταξης οικονομικών, ε, κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων και μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να οικοδομήσουμε με άλλους δωρητές και νέους φορείς που θα μπουν στην ανάπτυξη. Αντίστοιχα, η προετοιμασία για το πλαίσιο μετά το κοτονού μας επιτρέπει να επαναβεβαιώσουμε την στεναρή μας προσήλωση προς χώρες ΑΚΕ και ιδιαίτερα της Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα όφιλε ε, είναι, θα είναι στο κέντρο αυτών των ε, εξελίξεων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και τους εταίρους της παγκοσμίω. Πώς θα ε, διαμορφώσουμε, ε, θα, ε, τι θα σέψουμε την παγκοσμιοποίηση και πώς θα την αξιοποιήσουμε. Αυτή είναι η νέη στόχη μας. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, προσβλέπω πάρα πολύ συνεργασία μαζί σας για αυτές τις προτεραιότητες και παραπέρα θα αντλήσω ε, ε, πολλά διδάγματα από την παρούσα ακρόαση. Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη στην Ευρώπη που αναδεικνύει το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο και είναι προ όφελο και των εταίρων μας και των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ και πραγματικά προσβλέπω συνεργασία μαζί σας για αυτό το τόσο σημαντικό ε, θέμα που θα διαμορφώσει και τον κόσμο μας ολόκληρο τον πλανήτη για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστούμε κύριε Μιμίτσα. Να θυμίσω τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια. Σύμφωνα με τους κανόνες μας, εμείς τώρα θα συνεδριάσουμε και θα συντάξουμε επιστολή εξολόγησης. Δηλαδή θα γίνει αυτό και κλεισμένο το θύρον. Κυρία Πρόεδρε, μια παράκληση έχω μόνο. Ο, ο κύριος Ρούμπιχ ε, στο Twitter δεχόμαστε πολλά παράπονα ότι δεν παρακολουθούν την ακρόαση και δεν λειτουργεί σωστά το ίντερνετ στο κοινοβούλιο. Παρακαλώ να διορθωθεί για την επόμενη φορά. ναι. Ναι, υπήρξε ε, ένα μικρό πρόβλημα. Όσοι δεν είστε συντονιστές παρακαλώ να φύγετε από την αίθουσα και θα κάνουμε την αξιολόγηση, θα στείλουμε την επιστολή στους ε, Προέδρους των ε, Επιτροπών και μετά θα ληφθεί απόφαση ε, στην Ολομέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο το βράδυ, 6 ώρα, έχουμε άλλη ακρόαση. Δεν ξέρω γιατί η Επιτροπή μας έχει όλα τις, τα βραδινά ωράρια. Αύριο στις 6 και ευχαριστώ και τους Ιρμηνείς. Θα συνεχίσουμε σε λίγο.